Καλό για την ανοχή σας γιατί και εγώ έχω αποστείλει ε, επεξήγηση ψήφου που δεν έχει έρθει ακόμα στα χέρια σας. Βεβαίως κυρία Ντόιλ, χωρίς πρόβλημα θα δεχθούμε και τη δική σας. Επεξήγηση ψήφου λοιπόν τώρα. Ο κύριος Φατούτσο για την έκθεση Μπέλντερ και ένα λεπτό υπενθυμίζω αυστηρά. Signora Presidente, grazie. Eh, con grande piacere prendo la parola. Με μεγάλη ευχαρίστηση παίρνω το λόγο σε αυτή την τόσο σημαντική κοινοβουλευτική